Dear colleagues, please Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ πάρτε θέσεις. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε Uh, Θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με τις ψηφοφορίες. Το πρώτο σημείο είναι ο κανονισμός για τον υδράργυρο καταρρίξη της ε, οδηγίας ε, του κανονισμού συγγνώμη του 2008 μπορούμε να ξεκινήσουμε τη ψηφοφορία Mr. Ο κύριος Παολούτσι, Invite your assistant to... Στείλτε το βοηθό σας να φέρει την κάρτα σας. Και θα το λάβουμε υπόψη αυτό ότι προς τον παρόν δεν έχετε κάρτα. Εντάξει. Ωραία. 26 σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτονται. Δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά απορρίπτεται. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική υπαριθμών 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 187. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσανε όλοι. Καλά συμπαθάτε με κύριε Μπέλετ. Κύριε Πολίτη, έχετε την κάρτα σας. Πέρας. Κι άλλους κύριε Μπέντ, πέρα ψηφορίας. Απορρίπτονται. 189 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. 190 υπέρ. Α, όχι, συμπαθόταν. 191 και 192 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα συμβαστική παριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...214 της κυρίας Ριβαζή συμβατή με την ε, σύμβαση 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 231. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 237. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 236. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 235 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 239 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 240 υπέρ κατά απορρίπτονται. 241 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 242 υπέρ κατά απορρίπτεται 238 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 243 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 247. Και κόντρο. Τα αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Avete votato tutti il voto Paolucci. Paolucci ti γίνεται, ψηφίσετε. Il voto è chiuso. Per ψηφοφοριας ψηφοφορίας. 31-30. Και απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 248 με προφορική τροπολογία έχετε κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία όχι καλώς οπότε θα ψηφιστεί με την προφορική τροπολογία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, ήταν ε, ενιαίο. Δεν ήταν πρώτο τμήμα. Δέκα. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, έχει την κάτω ο κύριος Ντάντε. Και τώρα ψηφίζουμε την ε, τροπολογία 291. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 306. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 309 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το 310 είναι απαράδεκτο και ψηφίζουμε τώρα το 79 και το 313 που είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα όσον αφορά τα παραρτήματα καλύπτονται και άρα ψηφίζουμε τη συμβιβαστική Τι υπέρ. Κύριε Σόμερ, ξέρω ότι καθυστέρησα ε, να μιλήσω, αλλά την περασμένη εβδομάδα δεν μπόρεσα να είμαι παρούσα για τη συμβαστική εννέα Θέλω να πω ότι λέει ότι η δική μου ε, τροπολογία καλύπτεται, υποτίθεται. Θέλω να το πω για τα πρακτικά και ξέρω ότι δεν μπορώ να το αλλάξω επί της ουσίας να ψηφιστεί χωριστά. Θέλω να δηλώσω για τα πρακτικά ότι η συμβαστική εννέα δεν ε, περιλαμβάνει τη δική μου, γιατί λέει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλω να πω εγώ και να αλλάξω με την τροπολογία 341. Εγώ θέλω να δείξω ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικέ μεθόδους, ε, μέθοδοι συγγνώμη, και είναι πραγματικότητα κάπου και όχι face out για κάποιες ε, μεθόδους ε, παραγωγής και η συμβαστική λέει το αντίθετο. Παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά ότι η τροπολογία 341 δεν καλύπτεται από τη συμβαστική 9. Και παρακαλώ τους συναδέλφους τουλάχιστον της δικής μου ομάδας να καταψηφίσουν το συμβιβασμό. as you have uh, Όπως μας εξηγήσατε, ε, είναι αντίθετη η τροπολογία σας, οπότε εάν εγκριθεί η συμβιβαστική, τότε η δική σας τροπολογία σημαίνει ότι απορρίπτεται ή καταπίπτει. Τέλος πάντων, λαμβάνουμε υπόψη αυτό το οποίο μας εξηγήσατε. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Now we are going... Adesso andiamo alle... ai considerando e votiamo... Τώρα δίνουμε τις αιτιολογικές παραγράφους και ψηφίζουμε την 1.94 και 95 που είναι ταυτόσιμες. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, παραδείγμα 2, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97. Τροπολογία 97. Όμως ε, επειδή το 2 εγκρίθηκε καταπίπτει το 97. Πάμε στο 96. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα το 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 5 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Avete Ψήφισαν όλοι, πέρας. Α, εγκρίνεται. Votiamo adesso l'emendamento. Τώρα ψηφίζουμε το 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εμενταμέντο 6. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επτά. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές Εκατόν 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 8 υπέρ κατά εγκρίνεται 111 υπέρ κατά αποχές δέκα 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 115. Α, όχι, όχι. όχι. Καταπίπτουν γιατί το 114 εγκρίθηκε. Οπότε πάμε στο 10 του της του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα σε δύο τμήματα το 116. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 πόσο Ποιο? Α, το 127 του Μισελντοντέ Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα 140 του Μισελ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Avete votato tutti? Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 150 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158. Εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία. Έχετε κάποια ένσταση. Όχι. Οπότε το ψηφίζουμε με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 159. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, θα επαναλάβω την ψηφοφορία. Έτσι όπω ε, σηκώσατε τα χέρια, τα μισοσηκώσατε, δεν καταλαβαίνω τι έγινε. Υπέρ, κατά. Αποχέ, ε, ηλεκτρονικό έλεγχο. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ψηφίσατε όλοι. Mm. Πέρασε. It was difficult. Δύσκολο, δύσκολο ήταν. Και απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το 159 υπέρ. Κατά. Ποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Υπέρ για το 24 κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα η 25 σε δύο τμήματα. Πρώτον υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουν. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Voto finale sulla risoluzione legislativa. Η ψηφοφορία για το νομοθετικό κείμενο ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Ε, voto chiuso. Πέρασε. Approvato. Γκρίνεται. Adesso votiamo per eh, l'apertura del negoziato interistituzionale. Il voto. Ε, τώρα ψηφίζουμε όσον αφορά την έναρξη των ε, διοργανικών διαπραγματεύσεων. Ψηφίζουμε τώρα. Χρειάζονται 35 θετικέ ψήφοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. E λοιπόν, προχωρούμε. Και τώρα θα περάσουμε στην ψήφιση τη έκθεση. The vote is Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν τελειώσαμε ακόμα τι ψηφοφορίε. Έχουμε δουλειά ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι ψηφοφορία και αυτό. Είναι έκθεση Μπέρδε για το πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του λαθρεμπορίου αγρίων ειδών. Αρχίζουμε. Τροπολογία υπαριθμών 39. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 44 και 1 της ε, αλίας υπέρ. Ταυτίζονται αυτές οι δύο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα οι δύο, υπέρ, συμβαστική, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παρθμών 52 ψήφι, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 54 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 55 είπε. κατα Κατά. Αποχές εγκρίνεται. είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 56 ψηφί <coughs> Κατά αποχές Απορρίψεται. Η τροπολογία 79 και 126 μαζί. Υπέρ είναι ταυτόσιμες κατά αποχές απορρίπτονται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 68 που δεν καλύπτεται από το συμβιβασμό υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την 5 της Επιτροπής Αλίας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παρθμών 69. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ λέξεις. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 72. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 2 καταπίπτει. ΔΕΒΕ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε μία τροπολογία της αλίας. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία πες 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, συμβαστική 9, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 112 ε, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τώρα, είναι τα 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ πέρας. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη 14 της ΔΕΒΕ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 11. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 12. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 15. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. Ε, τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία 168. Ψηφί πέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ΔΕΒΕ 25 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 17 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Avete votato tutti? Ψηφίσετε άλλοι. The vote is Πέρας. Πάλι ισοψηφία. Respinto. Same votes. απορρίπτεται. Λυπάμαι πολύ. Αλλά δεν είναι σαφές. Έχουμε περίεργες πλειοψηφίες που διαμορφώνονται εδώ. Βεβαίως. Και πολύ. Πες τρία. Είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πού πάμε τώρα στην 182. Α, όχι, μόνο το πρώτο τμήμα θα ψηφίσουμε, για το δεύτερο καταπίπτει ή καλύπτεται. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ναι, το δεύτερο καταπίπτει. Τώρα θα ψηφίσουμε την 185. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 186, 187 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 Η τροπολογία τώρα 23, παρακαλώ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 26. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 27. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά mm. Συγγνώμη, μπορείτε να ξαναψηφίσετε 31 υπέρ παρακαλώ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. 32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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε ε, τη Γιούρι ε, ε, σε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε πολλές τροπολογίες της ΔΕΒΕ. Ας ψηφίσουμε όλες μαζί. Unblock. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται το αυτό για τις τροπολογίες Επιτροπής Γιούρη υπέρ όλων μαζί, κατά αποχές έλεγχος. Αβείτε... Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτονται. Και τώρα έχουμε πολλές τροπολογίες της Επιτροπής Αλίας, όλες μαζί και πάλι, υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Βασικά απορρίπτονται, αλλά τσεκ. Avete... Non avete votato tutti. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Υπάρχει κανείς που θέλει να ψηφίσει. Πέρας. Απερίφθησαν. Voto finale per voto elettronico. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται. Avete il voto è Πέρας. Εγκρίνεται Now we can go to the next. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Στην ημερήσια διάταξη ψηφίζουμε για τη γενική αναθεώρηση του στρικονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε εδώ μία ψηφοφορία για το, την, ε, για το συμβασμό 1β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ. Abbiamo Λοιπόν, τώρα έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση του συνάδελφου Μπουσόη για το αστικό δίκαιο και τη ρομποτική. Ψηφίζουμε επί του συμβασμού 1. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43. Τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία, ε, συμβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 66 υπέρ. 56 νομίζω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές να το τσεκάρουμε. Πέρας της εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 σε δύο μέρη το πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Και τώρα συμβιβασμός 6 για την παράγραφο 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60, 75, ε, συγγνώμη υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ. Τροπολογία 75. Mm. ναι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τώρα συνδυασμός υπαριθμών 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κύριε Ντάντι. Τροπολογία 91 σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε παρακαλώ το τρίτο μέρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100. Εδώ έχουμε προφορική τροπολογία. Είναι κανεί κατά τη προφορικής τροπολογία. Όχι. Λοιπόν, ψηφίζουμε επί τη 100 με την ε, προφορική. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 101. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 103. Υπέρ, κατά, απόχέ να το ελέγξουμε. ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογή, ε, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 120 σε τρία μέρη πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα συμβαστική λύση 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα τροπολογία 14 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος δε, καταπίπτει. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές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 αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Εγκρίνεται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. Συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή. Παρακαλώ, με άδελφοι. Όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε. Και όσοι δεν ενδιαφέρεστε για το επόμενο θέμα ή δεν θέλετε να λάβετε το λόγο. We wait one minute for giving the possibility. Ωραία, ας περιμένουμε ένα λεπτό για να μπορέσουν οι συνάδελφοι που θέλουν να αποχωρήσουν να το πράξουν. Dear colleagues, we can uh, start. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Παρακαλώ, οι διμερείς συζητήσεις εκτός της Επόμενο σημείο. Ανταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Καλέσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια βρήματα της μελέτης. Θα δώσω μέσα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εκπροσώπους. Τους δίνουμε μέσα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να παραστούμε σήμερα και να συζητήσουμε το πού κατέληξε αυτή τόσο σημαντική έκθεση. Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω ότι ο καθαρός αέρας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, για την υγεία μας και για το περιβάλλον και για την οικονομία. Ούτε χρειάζεται να τονίσουμε ότι δυστυχώς το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές ακριβώς λόγω της έλλειψης ποιοτικής ατμόσφαιρας στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ ψηλό. Μιλάμε για 400 χιλιάδες προώρους θανάτου ετησίω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό σαφώς είναι απαράδεκτο. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβαμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το τοπίο. Και γι' αυτό μετήλθαμε αυτή την οδηγία και έχουμε συγκέντρωση ε, των ε, μολυσματικών ουσιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπαμε ότι έχουμε καθεντήριες γραμμές από επιστημονική τεκμηρίωση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχουμε επομένω αυτές τις ε, κατευθυντήριες και πολλές φορές αυτές του ΠΟΗ είναι πιο αυστηρές διατάξεις αυτές που έχουμε εμείς θεσπίσει. Τώρα όσον αφορά τον ρυθμό υλοποίησης, αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει. Όσον αφορά τις οριακές τιμές που τάσει αυτή η οδηγία για τα κράτη-μέλη και ιδίω έχουμε τον ε, στόχο να συμμορφωθούμε προς ό,τι τάση η οδηγία μέχρι το 2020. Και σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσαμε να εργαστούμε εντατικά ούτως ώστε να υλοποιηθεί η οδηγία ταχύτερα βοηθώντας τα κράτη-μέλη για να μειώσουν την ε, μόλυνση του αέρα. Πάντως δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι ικανοποιητική και οδήγησε σε πάρα πολλέ ε, διαδικασίε και προσφυγέ επί παραβάση. Οπότε με λίγα λόγια έχουμε 29 τέτοιες ε, προσφυγές επί παραβάση για 19 κρατημέλη και 3 ρηπαντικέ ουσίε Να, μια εικόνα η οποία δεν είναι με τίποτα ικανοποιητική. Άρα δεν θα πρέπει να παίρνουμε αψήφιστα στο πόσες τέτοιε. Ε, αγωγές επί παρεμβάση έχουμε και υπάρχουν επομένως μεγάλα κενά στη συμμόρφωση τα οποία έχουν καταγραφεί. Ε, άρα γι' αυτό είπαμε τι χρειάζεται να κάνουμε τώρα. Πάντως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ε, αυτές οι προσφυγές ασκήθηκαν και ήταν θετική η απόκριση των κρατών μελών. Τους δώσαμε κίνητρα να βελτιώσουν την ε, ποιότητα της ατμόσφαιρας, ο πότων αέρα τέλος πάντων και Υπάρχουν τώρα τα σχετικά πλάνα, προγράμματα και σε τοπικό επίπεδο έχουν ε, ξεκινήσει κάποιες ε, πρωτοβουλίες. Όλο ένα και περισσότερες. Πάντως το τοπίο παραμένει πολύ ανεπαρκές. γιατί δεν είναι δυνατόν έτσι να ανταποκριθούμε στα στάνταρ που τάσει η οδηγία. Οπότε, για να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Όσον αφορά αυτές τις ε, παραβιάσεις για το PM10 έχουμε 16 κράτη-μέλη και σχεδόν όλα αυτά τα 16 κράτη-μέλη έχουν φτάσει στην φάση ε, στην αιτιολογημένη γνώμη και Πολωνία και Βουλγαρία ήδη έχουν παραπευθεί στο δικαστήριο γιατί έχουν τις χειρότερες επιδόσεις γιατί έχουν ξεφύγει πάρα πολύ όσον αφορά τις τιμές που προβλέπονται ε, άλλες ε, περιπτώσεις τέτοιων προσφυγών ε, έχει ανασταλεί η δίκασή τους και είπαμε επομένω ότι ε, έχουμε κάποιες περιπτώσεις για συγκεκριμένο διάστημα στο παρελθόν. Άρα τώρα τι κάνει το δικαστήριο, προσπαθεί να αξιολογήσει αυτή τη νέα προσέγγιση που δεν λαμβάνει υπόψη ε, την ε, ζημία που έχει γίνει, τι γίνεται με τις τιμές και επίσης γενικά ε, αξιολογεί τα μέτρα κατά αυτών των ρηπαντών. Και θα πρέπει όλες οι περιπτώσεις όμως όλες οι υποθέσεις αυτές να εξεταστούν και θα πρέπει επομένως να να, δούμε ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει γίνει, έχει διαπραχθεί η παραβίαση του δικαίου και τελικά δεν ε, επιβάλλονται κυρώσει, δεν εκδικάζονται περιπτώσει. Τώρα για την Βουλγαρία είπαμε τι έχει γίνει και αυτή η εκδίκαση έχει ανασταλεί γιατί θα πρέπει να εκδικαστεί η PM10 και μετά θα κυρώσει το δικαστήριο την νέα προσέγγιση. Έχουμε επίσης το διοξίδιο του αζότου και αυτό είναι ένας ρηπαντής. Η κατάσταση του Βασιλείου είναι πάρα πολύ σοβαρή. Έχουν υπάρξει πολλές καταγγελίες. Γι' αυτό και αυτό το είχαμε ως αφετηρία ενώ παρακολουθούσαμε τις άλλες υποθέσεις για τα άλλα κράτη-μέλη. Έχουν επίσης αρχίσει και έρευνες πιλωτικές όπου έχουμε υπέρβαση των οριακών τιμών και τώρα οι υποθέσεις που εξετάζουμε καλύπτουν 12 κράτη-μέλη και εκεί έχουν προσφυγές ή παραβάσει. είναι μια διατία. Και θα δούμε τι άλλο ενδεχομένως κάνουμε στο εγγύς μέλλον. αυτή η μόλυνση αφορά τα, τους διζελοκινητήρες στην πόλη. Έτσι έχουμε μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του αζότου. Τελευταίους μήνες έχουν γίνει μετρήσεις και έχουμε πάρα πολύ, πολλές μεγάλες πόλεις στα κράτη-μέλη που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μεγάλες υπερβάσεις. Μιλάμε για 100 πόλεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό. Οπότε για όλα αυτά προσπαθούμε να βάλουμε κάποιε προτεραιότητε, τι πιο σοβαρέ περιπτώσει, την έκθεση στου ε, ρηπαντέ σε σχέση με τον κόσμο στα κράτη-μέλη. Κοιτάμε πόσο έχουμε υπέρβαση οριακή τιμή, κοιτάμε πόσο κόσμο θίγεται και έτσι προσπαθούμε να έχουμε αντικειμενικό τρόπο τη κατάσταση. Όσο πιο πολύ είναι η μόλυνση, τόσο πιο αυστηρά θα πρέπει να είναι τα λαμβανόμενα μέτρα. Και σε σχέση με αυτό σας ξεκαθαρίζω το εξή. Όσον αφορά τις υπερβάσεις οριακών τιμών διοξιδίου του αζότου, δεν θέλουμε να δούμε ε, τι έγινε με, τα, με, τα, με, τις εκπομπές από αυτοκίνητα. Δεν θεωρούμε ότι αυτό θα, θα αρκέσει αυτές οι καινούργιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Φυσικά και τα αυτοκίνητα ρηπαίνουν πολύ περισσότερο από όσο θεωρητικά προβλέπεται. Άρα δεν μας αφορούν τα Euro Standards. Ε, γι' αυτό θέλουμε εμείς να διορθώσουμε με όλα αυτά τα οποία προτείνουμε στον συνομοθέτη όσον αφορά την έγκριση τύπου. Και είναι σαφές ότι από πλευράς περιβάλλοντος και από πλευράς ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και υλοποίηση αυτών ότι υπάρχουν μέτρα αποτελεσματικά και θα πρέπει να ληφθούν σχετικές αποφάσεις σε κάθε επίπεδο μέχρι και τοπικό όλα αυτά να εξεταστούν προσεκτικά και έτσι να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε προς τις οριακές τιμές για το διοξίδιο του αζότου. Υπάρχουν μέτρα τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν εξεταστεί πλήρως και αυτά είναι σημαντικά. Να, σας αναφέρω ενδεικτικά τι γίνεται με τη ζήτηση της μεταφορές, τις ε, ζώνες εκπομπών και εδώ υπάρχει πρόοδος, θέλουμε ακόμα περισσότερη ε, όσον αφορά κάποια μέτρα περιορισμού της κίνησης και κυκλοφορίας και εδώ σας τονίζω ότι έχουμε και τα τέλη και τους φόρους επί των καυσίμων και επίσης το πώς θα δώσουμε κίνητρα για αυτοκίνητα που εκπέμπουν λίγους ρήπαντες. Και εκεί που γίνει βήματα εργάζεται περισσότερη πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας διαβεβαιώνει. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυστηρά το τι γίνεται όσον αφορά την υλοποίηση και θα αξιοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε. Να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πλήρως την οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Θα πρέπει οποιαδήποτε περίοδος υπέρβασης γερακών τιμών να είναι όσο γίνεται πιο σύντομη. Τώρα όσον αφορά την έκθεση. Θεωρούμε πάρα πολύ θετικό το έργο το οποίο έγινε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και μεγάλη μας ικανοποίηση και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης συμπίπτουν με τις ε, ε, απόψεις της Επιτροπής. Και επομένω, ο εντοπισμός των προβλημάτων ε, υλοποίησης, hot spots και μας οδηγούν να δούμε τι αυστηρά μέτρα θα προηγηθούν σε κάθε επίπεδο για να υπάρξει συμμόρφωση με τους κανόνες. Ακριβώς όπως τα λέμε και εμείς στην έκθεσή μας. Είναι θέματα διακυβέρνησης, είναι θέματα συνέπειας λογικής των ε, εθνικών, τοπικών κλπ. μέτρων. Έτσι να βελτιώσουμε την κατάσταση. Όλα αυτά τα λέει και η μελέτη. Επίσης σας τονίζω ότι η μελέτη δεν είναι πάντοτε ακριβής. Σε ορισμένα σημεία παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που θα έπρεπε να επισημαθούν. Θα ήταν πιο καλή έτσι η μελέτη. Να, το κεφάλαιο το οποίο αφορά τις διαδικασίες των παραβάσεων, εκεί τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι τόσο σωστά. Μιλάμε τώρα για 19 και όχι 23 ε, κράτη-μέλη, 23 προσφυγές. Άλλα λέει η προσφυγή και άλλα, ε, συγγνώμη, άλλα μελέτη και άλλα ισχύουν. Επίσης έχουμε 10 δικαστικές αποφάσεις, 4 ανεκτέλεστες. Και αυτό ακριβώ γιατί έγινε η αλλαγή τη προσέγγιση και λοιπά και λοιπά, τα είπαμε προηγουμένως. Άλλο στοιχείο, η μελέτη επικεντρώνεται στην συμμόρφωση με τα πρότυπα, τα στάνταρ. Δεν λέει όμως για εποπτεία, για έλεγχο, όπως προβλέπει η οδηγία, που είναι πολύ σημαντικό. Και ε, το ίδιο φορά όσον αφορά, και το ίδιο ισχύει όσον αφορά το να αξιολογήσουμε την υλοποίηση. Επίσης, Θα σας τα πούμε, θα σας τα στείλουμε και εγγράφως. Δεν μπορώ τώρα να υψέθω σε όλες τις λεπτομέρειες. Επίσης, θα πρέπει να ολοκληρώσω πιο αισιόδοξα, γιατί όπως σας είπα, το τοπίο δεν είναι ικανοποιητικό, όπως το βλέπουμε εμείς. Και όσον αφορά την ε, υγεία των συμπολιτών μας και όσον αφορά το περιβάλλον. Άρα, οι πρόσφατες εξελίξεις μας κάνουν πιο αισιόδοξους. Τον Ιούνιο έκλεισε αυτή η προσωρινή συμφωνία για την οδηγία και αυτό δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν ήσασταν κι εσείς ως συνομοθέτες αποφασισμένοι. Και άρα ο πύχης θα πρέπει να παραμείνει ψηλά όπως τον έθεσε στην αρχή η Επιτροπή. Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που έγινε και είπαμε ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε κατά το ίμιση μείωση της ε, μόλυνσης του αέρα. Και όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν εάν και εσείς δεν ήσασταν δυναμικοί σε όλες τις συνομιλίες. Άρα θα πρέπει αυτή η πρόταση να εγκριθεί το συντομότερο και να προχωρήσουμε στη φάση της ε, υλοποίησης. Στη συνέχεια θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τα όσα τάση ο ΠΟΗ και τους στόχους μας του 50% δηλαδή το 2030 υπενθυμίζω, θα πρέπει να τα πάμε καλύτερα πρόθεσμα. Και επομένως θα πρέπει να φροντίσουμε για την ε, οδηγία IQ να εφαρμοστεί οπότε όπως και εσείς και εμείς θα κάνουμε ό,τι πάνε από το χέρι μας για να γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Για τις εξηγήσεις αυτές ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Γκερμπράντι; Julie first. Η Τζούλι Γκέρλινγκ, όχι ο κύριος Γκερμπράντι. Ναι, κάποια σχόλια θέλω να κάνω κι εγώ, μόνο. Σε σχέση με αυτή την αποτυχία, γιατί αποτυχία εγώ τη χαρακτηρίζω, επιβολής ε, της νομοθεσίας. Δεν είχα καμία πρόθεση να είμαι επικριτική. Τα εργαλεία και τα μέσα που διαθέτουμε είναι ακατάλληλα ή αποδεικνύονται ακατάλληλα όταν φτάνουν στα δικαστήρια. Ε, γιατί είναι τέτοιες οι καθυστερήσεις. Όταν μιλάτε εσείς για προσφυγές και διώξεις και μετά αμέσως για αναστολή, Καταλαβαίνω, βασικά δεν καταλαβαίνω γιατί νομικός δεν είμαι, δόξα τω Θεώ, ε, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα και κατανοώ γιατί γίνεται αυτό λόγω της νομοθεσίας η οποία χρειάζεται και ελέγχους και ε, ε, αντίβαρα αλλά για την ατμοσφαιρική ύπαρση δεν έχουμε χρόνο, την πολυτέλεια του χρόνου γιατί είναι πολύ χρονοβόρες αυτές οι διαδικασίες κάποια διαφορετική μέθοδο έχουν ε, υιοθετήσει οι πολίτες για το Ηνωμένο Βασίλειο να σας πω που κάπως το γνωρίζω έτσι λίγο σαν χώρα ε, για τι διώξεις πρέπει να συγχαρώ για να εκφράσω το θαυμασμό μου ε, σε οργανώσεις όπως είναι Client Earth που προσφέρουν κατά της κυβέρνησης και δεν είναι εύκολη υπόθεση γιατί είναι δύσκολο και το αγγλικό νομικό σύστημα η ένωμη τάξη μας δηλαδή για να μπορέσεις να πορευθείς και να φτάσεις. Και έχουν φτάσει και σε ε, ανώτατα δικαστήρια για την ατμοσφαιρική ρήπανση στο Λονδίνο. Μπορεί να έχει προχωρήσει η ζωή ε, σε βαθμό που οι πολίτες να έχουν ε, εγκαταλείψει την ιδέα ότι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα επιβάλλουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους στα κράτη-μέλη. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δουλειά για να βελτιώσει ορισμένα από τα δικαιώματα προσφυγής στη δικαιοσύνη παντού, έτσι, όχι μόνο για την ατμοσφαιρική ρήπαση, την ποιότητα του αέρα. Βλέπω μεγάλη προθυμία του Συμβουλίου να συζητάει τέτοια πράγματα και ουσιαστικά χρονοτριβή. αυτό θα πρέπει να έχει επιπτώσει, γιατί το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στι ανησυχίε των πολιτών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Το Συμβούλιο καμία βοήθεια και τα κράτη-μέλη το αυτό. Δεν ήταν ερώτηση βέβαια αυτό. Α, καταλήξω σε μια ερώτηση. Όταν οι δέσμοι μέτρων για την ποιότητα του ε, ατμοσφαιρικού αέρα ε, Πότε θα προχωρήσει, δεν θα το συζητήσουμε εδώ, να ξεφύγουμε από τον ΕΚ δηλαδή και να προχωρήσουμε στη νέα οδηγία. Προβλέπετε να γίνουν αλλαγές τα επόμενα χρόνια και μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θέλετε να βελτιώνετε, να βλέπετε να βελτιώνετε και με ποιο τρόπο μπορείτε να αναγκάσετε τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με μια νομοθεσία την οποία έχουν ε, δεσμευτεί να τηρήσουν. Φαίνεται ότι λησμονούν, έτσι. Δεν τους το έχουν επιβάλει εξωτερικά κανείς. Είναι μια υποχρέωση που έχουν αναλάβει εθελοντικά και από ό,τι φαίνεται δεν τηρείται. Προφανώ, γιατί ήρθατε εδώ για να μα πείτε ότι τα πάντα σχεδόν έχουν ανασταλεί και τι θα κάνετε εσεί γι' αυτό. Ο Γιάννη Γκερμπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά σκάνδαλα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει αυτό. Ο αέρας είναι κοινό αγαθό, είναι, ο καθαρός αέρας είναι θεμελιώδες δικαίωμα για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη και τι βλέπουμε. Ότι ακόμα και με μια σχετικά παλιά οδηγία, με προδιαγραφές πρότυπα που θα πρέπει να είναι πιο αυστηρά, τα κράτη-μέλη αρνούνται να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, τι απαραίτητε αποφάσεις για να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και για μένα συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν είναι ο ίστατος στόχος. Ο στόχος είναι να αγγιηθούμε πιο καθαρό αέρα. Δεν είπα καθαρό αέρα, είπα λίγο πιο καθαρό αέρα. Αναφερθήκατε σε 29 παραβιάσει σε 19 κράτη-μέλη. Η δική μα μελέτη του Κοινοβουλίου ε, νωρίτερα φέτο, αναφέρεται σε παραβιάσεις, ε, διαδικασίες σε παραβάση μάλλον κατά 23 κρατών, κρατών μελών. Εάν αυτό δεν αποδεικνύει την αποτυχία του ευρωπαϊκού συστήματος, τι να πω. Λοιπόν, το έχουμε πάρει πολύ ελαφρά την καρδία το ζήτημα αυτό ως Κοινοβούλιο, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Έχω κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τον επόμενο μήνα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια για την τελική συμφωνία σχετικά με την οδηγία ΝΕΚ. Εγώ θα ψηφίσω κατά αυτής της συμφωνίας. Σας το λέω από τώρα, συγγνώμη. Τζούντι, αλλά έτσι είναι. Διότι δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη. Εσύ πιστεύεις ότι είναι παρκές αυτό, ότι αρκεί. Επίσης ε, Πιστεύεις ότι η αναθεώρηση ε, της οδηγίας από ηθικής πλευράς, από πολιτικής πλευράς είναι απαραίτητη. εντάξει, φυσικά και είναι, αλλά δεν τολμάτε να το κάνετε. Διότι τα κράτη-μέλη προσπαθούν ήδη την παρούσα οδηγία να την παρακάμψουν. Τρίτον, ακούω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με τα δεδομένα που έχουν ε, συλλεχθεί στα κράτη-μέλη. Ακόμα και η πόλη των Βρυξελών δεν συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα. Η Ρίντο Λαλουά από ό,τι μου είπαν, όπου όλοι ερχόμαστε υπερβολικά συχνά, έκλεισε τα σημεία μέτρησης, διότι ξέρουν από τον προτέρων ότι δεν πρόκειται να πληρούν τις προδιαγραφές. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο λοιπόν για την ε, αξιοπιστία των δεδομένων στα κράτη-μέλη. Και κάτι ακόμα επειδή έχω ασχοληθεί και με το Dieselgate, είπατε ότι το μεγάλο πρόβλημα στις ευρωπαϊκές πόλεις είναι τα diesel. Τώρα έχουμε αυτή την ε, τρομακτική απόφαση ε, για τους παράγοντες σχετικά με τα οχήματα για τα κριτήρια συμβατότητας. Η κυρία Ντάλι. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν που ήρθε εδώ σήμερα και μας έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα εδώ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε πλήρη επικυροποιημένα στοιχεία για όλες τις πηγές ρήπανσης για να φτάσουμε στις κατάλληλες πολιτικές ε, που να μπορούν να κάνουν τη διαφορά, χρειαζόμαστε αυτά τα πλήρη επικαιροποιημένα στοιχεία. Όταν λοιπόν έχουμε την ανησυχία ότι αυτές οι πληροφορίες δεν μας δίνουν την ε, ε ακριβή εικόνα, μπορούμε να οδηγηθούμε σε πολιτικές αποφάσεις που δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς μπορούμε τελικά να έχουμε τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία για να πάρουμε αποφάσεις ε, απαραίτητες. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι τα κατόφλια ε, για τα συγκεκριμένες ουσίες ε, έχουν ξεπεραστεί σε πολλά κράτη-μέλη. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει την υγεία των συμπολιτών μας. Και τα κράτη-μέλη για άλλη μια φορά κολυσιεργούν για πολλές σημαντικές νομοθεσίες που μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά ε, στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Ο κ. Γκερμπράντι προηγουμένως αναφέρθηκε και στις εκπομπές των οχημάτων ε, και αυτό μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά ε, και αυτό επηρεάζει την υγεία των συμπολιτών μας. Ανησυχούμε λοιπόν με τις πληροφορίες αυτές ότι εδώ γίνεται μια απόπειρα να νερωθεί το τρίτο πακέτο RDE και αυτό λοιπόν μας ανησυχεί. Αντιλαμβανόμαστε και πιστεύουμε ότι η διαχείριση της ποιότητας ε, του αέρα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική πολιτική και βεβαίως πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία μέσα των διαφορών υπηρεσιών που συμμετέχουν στο σύστημα αυτό έτσι ώστε όντως οι προληπόμενες δράσεις να ολοκληρωθούν για να μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, βεβαίω η ΝΑΚ είναι μια πολύ, ένα πολύ σημαντικό βήμα καθώς και η εισαγωγή των βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών και της καλύτερης διαθέσιμης πρωτο, ε, ε, τεχνολογίας, ε, τα οχήματα μεταφορών τα οποία είναι ενεργειακά καθαρά. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που πρέπει όμως να πιέσουμε ως ε, Κομισιόν αλλά και ως και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να σταματήσουν να κολλησιεργούν τα κράτη-μέλη. Διότι εάν δεν πάρουμε στα σοβαρά την ποιότητα του αέρα θα ερχόμαστε εδώ ξανά χρόνο με το χρόνο να μιλάμε για τις εκπομπές και να μιλάμε για διαδικασίες σε παραβάση κατά κρατών μελών ενώ στην πραγματικότητα η την άμεση αρνητική επίπτωση τη βιώνουν οι συμπολίτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σεκχάουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το όσα μας είπε. Πολλά είπαν για τη σημασία του να έχουμε καθαρό αέρα έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελα να τονίσω κάτι ε, που έχουμε με ε, τέτοιες πολιτικές ε, κάθε φορά που συζητούμε την οδηγία αυτή Όλοι κοιτάνε στα κράτη-μέλη ε, και όταν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τη δουλειά τους απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενεργοποιεί τις διαδικασίες. Αλλά κάθε φορά που συζητούμε κάποιες ε, ε, πολιτικές από την αρχή ακούμε διάφορες ε, φωνές, ε, λόμπι, ε, που μας λένε ναι, ναι, ναι, να καθαρίσουμε τον αέρα, αλλά όχι εμείς, κάποιος άλλος κλάδος που ρηπαίνει περισσότερο. Εκεί θα πρέπει να το δούμε στην πηγή, δηλαδή ο ρηπαίνων ποιος είναι κάθε φορά και ο ρήπος και ο ρηπαντής. Ας πούμε πάμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία δεν συμμορφώνεται και δεν τα τηρεί. Παράδειγμα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν το έχουμε αντιμετωπίσει στη ρίζα του το κακό και στην πηγή της ρήπανσης. Ε, θέλω να ρωτήσω λοιπόν κάτι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Τώρα έχουμε για ε, τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, έχουμε ε, μια διαδικασία, αλλά ψάχνουμε να βρούμε τις ναι. βέλτισες τεχνικές, ε, δηλαδή να ε, έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και συμπαραγωγή και τα λοιπά. Είναι κάπως θολό το τοπίο εκεί. Έτσι θα καθαρίσουμε τον αέρα μας. Θα πρέπει να καθαρίσουμε τις πηγές της ρήπανσης. Αυτό είναι για μένα και ε, έχω την αίσθηση ότι αυτό καθυστερεί πολλές φορές και είναι κρίσιμο. Και πολλές φορές ή καμιά φορά μάλλον ακούω ότι επειδή είναι τόσο μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλύτερη, η βέλτιστη τεχνική δεν είναι τόσο προηγμένη όπως το παρελθόν, δηλαδή πάει στην άλλη κατεύθυνση. Τι είναι αυτό, δηλαδή στις τεχνικές μας εμείς χειροτερεύουμε, γελία πράγματα είναι αυτά. Θέλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κοιτάξει αυτό και να δούμε και να φροντίσουμε να προοδεύουν οι τεχνικές και όχι να επιδεινώνονται. Έχω και άλλη ερώτηση, ε, την ίδια με τον κύριο Χερμπράντη. Δηλαδή, πόσο βέβαιοι είμαστε ότι τα κράτη-μέλη μετρούν με το σωστό τρόπο τους ρήπους. Δηλαδή, αν γίνουν οι μετρήσεις στα σωστά σημεία και δεν είμαστε πολύ κριτικοί στις προβολές, υπάρχει και άλλη ατμοσφαιρική ρήπανση που δεν τη βλέπουμε, που δεν τη μετράμε. Πώς είμαστε βέβαιοι ε, ε, για την πραγματική ποιότητα το ατμοσφαιρικό αέρα. Και όλες οι Βρυξέλλες ε, είναι ε, κρίσιμες αν έρχεσαι με ποδήλατο το πρωί και η Χουίντελα βεβαίως, να εκεί να μετρήσουμε. Δεν θα πάμε σε κανάλι λιβάδι να μετράμε την ατμοσφαιρική ρήπαση. Also we will vote against the NEC direct... Και η κυρία Γκέρλινγκ τα ξέρει αυτά. Εγώ καταψήφισα την, την ε, οδηγία ΝΕΚ για τις ε, οροφές εθνικών εκδοχών. Υπάρχουν πολλά λόμπι και της γεωργίας. Για να εξαιρούνται κάποιες πηγές ρήπανσης. Και ο αέρα μας παραμένει ε, βρώμικος. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, βέβαια και όλοι εδώ στην Επιτροπή μας θέλουμε να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Πάντα παρουσιάζει ενδιαφέρον να ακούμε απόψεις ε, και αναλύσεις από πλευράς κομισιών. Και οι υποφαινόμενοι, ξέρετε, επί 17 έτη ήμουν επικεφαλής ενός συμβουλίου που ε, ήλεγχε την ποιότητα του αέρα στην περιφερειά από το 1990 μέχρι το 2008 και ξέρω το θέμα. Βέβαια ότι καταβάλλονται κάποιες ε, προσπάθειες, οπότε, όποτε κάτι αποφασίζουμε και υπάρχουν κάποια αποτελέσματα κάποια στιγμή τελικά, έπαιρνε ε, πάρα πολύ καιρός γιατί έχουμε το θέμα του τι γίνεται από τις μεταφορές, τι γίνεται στις, πόλεις, τι γίνεται στις αστικές περιοχές, άρα θα πρέπει να δούμε πώς πρέπει καλής να νομοθετεί. Ε, φυσικά και το θέμα του τι θέλει ο κόσμος. Ε, πολλές φορές δηλαδή δημιουργούμε προβλήματα για την ε, κυκλοφορία αυτοκινήτων, οπότε αυτά είναι δυσάρεστα για τον κόσμο. Έχουμε επίσης και το θέμα της ε, θέρμανσης τη πόλη. άρα πρέπει να βελτιωθεί η τεχνολογία. Και στην αυτοκινητοβιομηχανία έχουμε την ΙΜΗ στην Εξεταστική Επιτροπή μας και γνωρίζουμε τι σκάνδαλο ξέσπασε σε σχέση με την Volkswagen, η οποία τώρα θα πρέπει να κάνει μια στροφή 180 μοιρών. επίση ε, θα πρέπει τώρα να υποχρεώσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία να ελέγξει κάποιες λύσεις πιο ποδοτικές από ό,τι ή μέχρι σήμερα. Αυτό ε, μας κάνει σκεφτούμε ότι καλές είναι και ακυρώσει, αλλά καλύτερα είναι τα κίνητρα. Άρα θα πρέπει να παρακινήσουμε όλους να καταβάλουν προσπάθεια. Τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, τη βιομηχανία γενικότερα. Γιατί είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ε, η θέρμανση στις πόλεις, οι τοπικές αρχές. Δεν είναι για μένα το καλύτερο η επιβολή ποινών και κυρώσεων. γιατί έτσι έτσι και έχουν λίγα χρήματα οι τοπικές αρχές, αλλά θα έπρεπε ε, ε, τους σχετικούς πόρους να τους κατευθύνουμε προς την παροχή κινήτρων. Άρα να τα δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Ναι, έχουμε βήματα προς τα μπρος. Έχουμε κάνει, αλλά θα πρέπει να βρούμε και τα σωστά μέσα για να παροτρύνουμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Ευχαριστώ κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να λάβω το λόγο, ούτω ώστε να σας πω όσον αφορά την κατάσταση ότι είναι πολύ περίπλοκη, πολύ μπερδεμένη. Και αυτό προκύπτει κάθε φορά που κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και τελικά δεν βλέπουμε κανένα πιο αποτέλεσμα. Και με εντυπωσίαση η διαφορά μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχέση με τις προσφυγές επί κατά των κρατών μελών. Αυτή η διαδικασία ξεκινά βέβαια από την Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον. Όμως τελικά έχουμε αδράνεια, τέλος πάντων έλλειψη ε, πρωτοβουλίας από τις άλλες συναρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Να, τι πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο προκύπτει από τον Dieselgate και την Ελληνική Επιτροπή. Όλοι πια έχουν καταλάβει το τι γίνεται όσον αφορά το πόσο λίγο ρεαλιστικές είναι οι σχετικές προδιαγραφές και οι κανόνες. Το, το Και Είδαμε πώς πιστοποιούνται τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, επιτήρηση στην αγορά. Μου φαίνεται απίστευτο ότι τόσα χρόνια δεν υπήρχε κάποιο είδου ε, πυγμή ούτως ώστε εγκαίρως να έχουν θωρακιστεί οι σχετικές δοκιμές. Από το 2007 τα ξέρανε οι βιομηχανίες, δηλαδή 8 χρόνια πριν. 8 χρόνια από τότε που υπάρχει το Euro 6 σαν στάνταρ. Ξέραν ότι οι ορικές τιμές δεν τηρούνται. Ε, να όμως παρόλα αυτά και φέτος προσπαθούμε να υιοθετήσουμε το χιλιοστό, τον ιωστό μέτρο για, ε, για αυτού του είδους τα περιβαλλοντικά στάνταρ. Και κάνουμε και τα στραβά μάτια σε όλους αυτούς οι οποίοι ακόμα και σήμερα δεν σέβονται τις ωραϊκές τιμές. Στους διζελοκινητήρες. Άρα, θα πρέπει και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει κάποιο είδου δυναμική ε, πρωτοβουλία, αλλά και από τα κράτη-μέλη, το έχουμε ξαναπεί. Και μια τελευταία μου σκέψη. Πώς συμβιβάζονται, πώς, πώς ταιριάζει το ότι έχουμε τις ε, παραβιάσεις σχετικέ με τον ατμοσφαιρικό αέρα και από την άλλη μεριά δεν έχουμε κάποια μέσα, κάποια εργαλεία σαν τοπικές αρχές ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή την ε, μόλυνση και ρήπανση του αέρα. Έχουμε το, το, το Euro 6 ή αλλά κάτι πιο, πιο αυστηρό, τόσο να τηρηθούν οι οριακέ τιμέ για τα αυτοκίνητα. Γιατί μια τέτοια χολή διαδικασία παραβίαση που φαίνεται ότι δεν κάνει τίποτα. Έχουμε τι τοπικές αρχές, τι περιφερειακές αρχές, αυτοί θα έπρεπε σοβαρό τρόπο να έχουν δράσει. Άρα αυτό είναι μια αντίφαση. Και τέλος, σας υπενθυμίζω ότι ανησυχεί ο κόσμος τόσο πολύ που συνέχεια έρχονται εδώ αναφορές. Ε, πάρα πολλές στην Επιτροπή των αναφορών έρχονται από χιλιάδες Ευρωπαίους. Και όλοι αυτοί διψούν για μία απάντηση. Ε, αυτό φυσικά και μας τονίζει το πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα νομίζω ότι θέλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Ε, θα απαντήσω σε κάποιε ερωτήσει. Θα δώσω το λόγο και στον συνάδελφο Γιόν Κοντέσκου, ο οποίο είναι αυτό που παρακολουθεί τι ε, παραβάσει, τι διαδικασίε επί παραβάσει, θα σχολιάσει κυρίω το ερώτημα τη κυρία Γκέρλινγκ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω ανάποδα με τα τελευταία ερωτήματα που τέθηκαν. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τι ε, παραβάσει που έχουν ξεκινήσει, τι διαδικασίε που έχουν ξεκινήσει σε σχέση με τη Γενική Διεύθυνση Grow, όπω ξέρετε η κυρία Μπιανκόφσκα, έκανε κάποιε αναφορέ, στι διαδικασίε στις ε, ε, διαδικασίες και παραβάσεις όταν πήγε στην Επιτροπή, αλλά δεν θα σχολιάσω, εξετάζεται πάντως το θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτά που είπε η κυρία Εύγε για τον τύπο έγκριση το γεγονό ότι δεν είναι αποτελεσματικό το σύστημα. Είναι αλήθεια ότι είναι αποτελεσματικό. Γι' αυτό και η Κομισιόν στι 27 Ιανουαρίου πρότεινε να διορθωθεί σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου. Και πρέπει να πω ότι όταν βλέπω τι προκύπτει από τι εργασίε του Κοινοβουλίου επ' αυτού, είδα την πρώτη εκδοχή τη έκθεση και σίγουρα υπάρχουν λόγια ανησυχία, διότι πολλά από τα μέτρα εποπτεία τη αγορά που έχει προτείνει η Κομισιόν εξετάζονται επιφυλακτικά, τουλάχιστον από πλευρά εισηγητή. Οπότε εμά μα απασχολεί αυτό, να νερωθεί δηλαδή η πρότασή μα. Σε ό,τι αφορά τώρα την έλλειψη περιθωρίου ελιγμών για τις τοπικές αρχές να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την μόλυνση τη ατμόσφαιρας. Ε, είναι περίπλοκο το θέμα αυτό, έτσι. Πολλά μπορούν να γίνουν σε τοπικό επίπεδο και πολλά από αυτά φέρνουν αποτελέσματα. Αναφέρθηκα προηγουμένως στις ζώνες χαμηλών εκπομπών, τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που παίρνονται σίγουρα οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω και η μελέτη σα προ αυτήν την κατεύθυνση πάει. Έχουμε στοιχεία δηλαδή τα οποία δείχνουν ότι αυτό ο, ο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό όμω που είναι επίση είναι σαφέ είναι ότι αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε ε, και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο υποστήριξη. Και αν δούμε τα κίνητρα που έχουν δοθεί τα φορολογικά τα τελευταία χρόνια για τα αυτοκίνητα diesel, ε, εδώ υπάρχει μια αντίφαση σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει και σίγουρα δεν βοηθούμε έτσι το έργο των τοπικών κοινωνιών. Το λέω αυτό για να πω ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα σε τοπικό επίπεδο, μπορούμε να πάμε πέρα από αυτά που έχουν γίνει ε, σε διάφορους δήμους της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της παρακολούθηση τη εποπτείας, ε, τότε το έθεσαν ε, πολλοί από εσά. Εδώ σίγουρα τα πράγματα δεν είναι τόσο θολά ε, όσο φαίνονται. υπάρχουν σοβαρές ε, προδιαγραφές για τα δείγματα που πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά, που πρέπει να προέρχονται από τις περιοχές όπου, έχουν, έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Εντάξει, δεν είναι βέβαια συνολικό, είναι αντιπροσωπευτικό δεν είναι εξαντλητικό. Μπορούμε όμως να αποκτήσουμε μια εικόνα ε, του μεγέθους του προβλήματος, της κλίμακας. Μπορεί για σας αυτό να, να μην πηγαίνει αρκετά μακριά. Δεν έχουμε δηλαδή δυνατότητα επιθεώρησης εμείς για να δούμε λεπτομερώς πώς αυτό εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Πρέπει δηλαδή να βασιστούμε στις πληροφορίες που μας δίνουν. Έτσι λειτουργεί το σύστημα υπάρχουν κάποιες απαιτήσει στην νομοθεσία που δίνουν εγγύησει ότι αυτό που ε, ε, έχουμε ε, ακολουθεί τη σωστή οδό, στον δρόμο, αυτό που συμβαίνει, εν πάση Κάτι άλλο που αναφέρθηκε προηγουμένω, αναφέρθηκε συχνά. Όντω, θα πρέπει να εξετάσουμε όλε τι πηγέ. Δίνεται μεγάλη έμφαση και πολύ σωστά στα δίζελ, στις οδικές μεταφορές, στην ε, οδική κυκλοφορία, ιδιαίτερα μετά το, το σκάνδαλο του Dieselgate. Όμως ε, υπάρχει και το θέμα της ε, θέρμανσης, της οικιακής. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε άλλες εκπομπές μεταφορών, τα, στον IMO θα γίνουν συζητήσεις για μια πιθανότητα ανώτατου ορίου ε, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές ε, τις ε, θαλάσσιες. Ε, είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει. Τώρα, κατά πόσο πάμε αρκετά μακριά, κατά πόσο είμαστε όμοιροι κάποιων λόμπι, για αναφορά και στην οδηγία ΝΕΚ, ακούστε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρότασή μας θεωρούμε ότι ήταν η, η πιο σωστή και για την αμμονία και για τη μεθαΐνη, ε, το μεθάνιο, συγγνώμη. Εμείς συγκροθούμε να θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση πρέπει να υποστηριχθεί διότι θα βελτιώσει την κατάσταση. Θεωρούμε λοιπόν ότι σίγουρα αυτό θα αποτελέσει σημαντική βελτίωση. Δεν είναι βεβαίως μια βελτίωση η οποία ε, ανταποκρίνεται στην αρχική μας φιλοδοξία, αλλά ε, είναι μια ε, νομοθεσία που σίγουρα βελτιώνει τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημά σας για το LCP, το σημείο, το σημείο, το σημείο LCP και τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα, ξέρω ότι μια σειρά από παράγοντες μα ε, επικρίνουν, μας επικρίνουν για το επίπεδο φιλοδοξίας θα πρέπει να το δω το θέμα για να απαντήσω πλήρω. Ε, είμαστε στη φάση ολοκλήρωση ε, σε επίπεδο κομισιών για να μπορέσουμε να έχουμε ε, έναν αντίκτυπο σημαντικό και για την υγεία και το περιβάλλον. Αυτό είναι ο στόχος μας, να εγγυηθούμε ότι θα είναι επαρκώς φιλόδοξο το όλο εγχείρημα και αυτό που είπατε για το BAT, το οποίο τελικά θα ευθυγραμμιστεί με τον κατώτερο κοινό παρονομαστή. Εμεί δεν το βλέπουμε έτσι το θέμα των BAT ε, στην ε, Κομισιόν, στην δική μου ε, γενική διεύθυνση. Δεν κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της αναθεώρησης για την ποιότητα του αέρα και τη σχετική οδηγία, το 2013 όταν προετοιμάσαμε το πρόγραμμα για το καθαρό, το καθαρό αέρα είχαμε αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται να θεωρηθεί οδηγία. Είχαμε πει πρέπει να ε, επικεντρωθούμε, να επικεντρώσουμε στις προσπάθειές μας να φτάσουμε σε, σε μια πλήρη εφαρμογή το 2020. Αυτός είναι ο πολιτικός στόχος τον οποίο είχαμε τότε. Είναι σαφές στο πλαίσιο ε, της, του κύκλου αναθεωρήσεων ε, θα φτάσουμε, θα φτάσουμε ξανά, θα το βρούμε μπροστά μας το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται εμείς να κρυφτούμε σε καμιά περίπτωση θα πρέπει να δούμε τις εξ, εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ε, ιδιαίτερα ε, σε επιστημονικό επίπεδο, σε επίπεδο νέων ε, στοιχείων, νέων γνώσεων που έχουμε. Έχει εργαστεί από αυτού περαιτέρω και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια του τακτικού fitness check που αφορά και τι λοιπέ νομοθεσίε, είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Θα δούμε δηλαδή κατά πόσο μπορεί να φτάσουμε σε μια ευθυγράμμιση με τι κατευθύνσει γραμμέ τη Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία, που είναι κάπω πιο φιλόδοξα από τι δικέ μα, σε αφορά τα πρότυπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα τεθεί επιτάπητο όταν θα εξετάσουμε την αναθεώρηση. Για το θέμα των παραγόντων συμμόρφωση που, που επιλέχθηκαν με βάση το πακέτο RD2. Ε, το ρώτησε ο κ. για το πώς είμαστε ικανοποιημένοι. Ακούστε, εμεί θα προτιμούσαμε να πάμε πιο μακριά. Ε, σε κάποιες περιοχές του κόσμου, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει καν τέτοιο πράγμα, έτσι, παράγοντες ε, συμβατότητας. Ε, τώρα, αυτό το πακέτο ε, αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το παρελθόν. Είναι μια βελτίωση. εντάξει, ίσως να μην πάει όσο μακριά θα θέλαμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα γίνει και υπάρχει μια, υπάρχει μια έδρα σε αυτό το ε, σύστημα που μας επιτρέπει να προβούμε σε βελτιώσεις. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια βελτίωση, θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο φιλόδοξοι. Ο Επιτροπός μου ήταν σίγουρα πιο φιλόδοξος αρχικά στις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να σας κάλυψα έγινε αναφορά στους πολίτες που οθούν για αλλαγές ε, και τις διάφορες ε, ε, νομικές διανέξεις που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο, αυτό που συμβαίνει στο Μένο Βασίλειο με το Client Earth μπορεί να μην ισχύει αλλού. Έτσι, η κινητοποίηση και το κατά πόσο είναι κάτι αυθεντικό που έρχεται προς τα κάτω δεν ισχύει παντού. Σε κάποιες χώρες ενδεχομένως είναι πιο δύσκολο δηλαδή να βασιστούμε σε τέτοιου κινήματα. Ε, αυτές ε, οι δράσεις βεβαίως πάνε χέρι-χέρι. Ε, έχουμε κάποια καλά νέα από περιφερειακές, εθνικές υποθέσεις στα δικαστήρια. Ιδιαίτερα στις 14 Σεπτεμβρίου στο Ντίσσελντροφ στη Γερμανία ε, υπήρξε μια υπόθεση όπου καταλήξαμε ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερες δράσεις σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο για να περιοριστεί κυκλοφορία σε κάποιες περιοχές έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι ε, περί, και, και οι τιμές που προβλέπονται ε, για την ποιότητα του αέρα και τη σχετική οδηγία. Πολλά λοιπόν έχουν, μένουν να γίνουν, αλλά σίγουρα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει πράγματα και μέσω της διαδικασίας παραβάσης θέλουμε και ένα μήνυμα για το επίπεδο πίεσης το οποίο είναι ορατό για τα κράτη-μέλη και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Δίνουμε δηλαδή κίνητρα για να παρθούν αποφάσει πάνω προ την κατεύθυνση. Μπορεί να μην αρκεί, αλλά είναι μια προσπάθεια. Και τώρα δίνω το λόγο στον συνάδελφο. Πριν περάσουμε στα νομικά ζητήματα, μια συμπληρωματική ερώτηση, κύριο Σεκχάουτ. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι τα μπάτσι, τα LCP θα ενισχυθούν Είπατε ότι δεν θα χαθούν, δεν ζήτησα εγώ τέτοιο πράγμα. Υπάρχει κίνδυνος να παραμένουν στο ίδιο επίπεδο ή να χαλαρώσουν κάπω. Αυτό σας ρώτησα. Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι θα είναι αυστηρότερα τα κριτήρια αυτά. Όπως σας είπα, δεν παρακολουθώ αυτό το θέμα άμεσα. Θα πρέπει να δω ποιες είναι οι ε, τελευταίες εξελίξεις για να σας απαντήσω. Αυτά που σας είπα ισχύουν. Το επίπεδο φιλοδοξίας που έχουμε επιδείξει ε, θέλουμε να διατηρηθεί. Δεν παρακολουθώ τη συζήτηση αυτή, επαναλαμβάνω στενά. Βλέπω όμως να διονται διάφορα ζητήματα. Θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή από κάθε σκοπιά. Βεβαίως ε, θα παραμείνουμε σε αυτή μας τη φιλοδοξία και σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος και σαφής όσο γίνεται για τα νομικά ζητήματα. Αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ περίπλοκες και όπως γνωρίζετε στο παρελθόν ε, και στείλαμε τέσσερις ε, υποθέσεις ε, στο δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ε, ελήφθησαν και αποφάσεις κατά των κρατών. Ε, αυτό ήταν ένα είδος fast track γιατί τα κράτη-μέλη υπερεύσαν τα όρια. Αποφάσεις έχουν εκδοθεί, αλλά δυστυχώς ε, ήταν περιορισμένες χρονικά στο παρελθόν και δεν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια. Ήταν για την περίοδο 2004-2007. Τώρα πώς να βελτιώσουν τα κράτη-μέλη κάτι που συνέβη στο παρελθόν. Είναι τελεσμένο. Ε, σταματήσαμε λοιπόν και αναθεωρήσαμε τη στάση μας και την προσέγγισή μας. Αρχίσαμε νέα δράση. Πάντα θα υπάρχει μια χρονική υστέρηση. Ε, μέχρι να φτάσει στο δικαστήριο μια υπόθεση, τα στοιχεία που έχουμε είναι παλαιότερα. Και το, συμβούλιο, συγγνώμη, το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί επί που ε, είναι του παρελθόντος για την τελευταία περίοδο, το τελευταίο έτος ας πούμε, δεν έχουμε στοιχεία για τα οποία θα πρέπει να ε, εξεταστούν και να κυρωθούν, να εγκριθούν από τα κράτη-μέλη. Για να πιστεί λοιπόν το δικαστήριο να δώσει λύση, τι κάναμε. Αρχίσαμε να ε, προσφεύγουμε ε, όταν υπάρχει σοβαρή και επίμονη ε, αποτυχία, όταν δεν βελτιώνεται η κατάσταση σε ένα ε, βραχή διάστημα και επιμένουν αυτά. Και επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρχίσαμε να στοχεύουμε και την έλλειψη καταλήλων μέτρων βάσει του άρθρου 23 της Οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Είναι πολύ βαριά όμως αυτή η διαδικασία. Ε, σε σχέση με την προηγούμενη ταχεία, γιατί χρειάζεται ανάλυση μέτρων και αυτό καλύπτει εκατοντάδες περιοχών, ζωνών λοιπά Και πρέπει να πιστεί το δικαστήριο ότι τελικά είναι κατάλληλα τα μέτρα και για να αλλάξει ε, την απόφαση. Και καμιά φορά, και καμιά φορά πολύ συχνά τα κράτη-μέλη λαμβάνουν ε, τελευταία στιγμή τέτοια μέτρα Και δεν μπορούμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο εναντίον ενός μέτρου που ακόμα δεν έχει ε, αρκετή ζωή για να αποδείξει την ε, χρησιμότητά του και την αποτελεσματικότητά του. Και πραγματικά καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια, τεράστια. Και θέλουμε να δούμε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις της Βουλγαρίας και της Πολωνίας. Για τη Βουλγαρία, μάλλον αρχές του 2017 θα έρθει η απόφαση πριν τα τέλη του έτους δεν αναμένεται. Ε, αν η προσέγγιση μας λοιπόν επιβεβαιωθεί, τότε οι υπόλοιπε υποθέσεις που δεν έχουν ε, ανασταλεί θα προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Και τώρα συζητούμε για το PM10, PM10 και προσπαθούμε να διατηρήσουμε την πίεση, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, στα κράτη-μέλη. Ούτε έχουν κλείσει, ούτε έχουν ε, εγκαταληφθεί. Ε, συνεχίζεται αυτή η προσφυγή επί παραλήψη. Έχουμε 12 περιπτώσεις υποθέσεις συνολικά. Οι συγκεκριμένες είναι στο στάδιο της αιτιολογικής, ε, αιτιολογημένης μάλλον. Είναι πολύ περίπλοκα τα θέματα. Άλλο σημαντικό ζήτημα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τη δράση που λαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο και τη θεωρούμε συμπληρωματική προς τη δική μας. Είμαστε σε στενή επαφή με τις ΜΚΟ, Client Earth και και βεβαίως θέλουμε να βελτιωθεί και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε κάποια κρατημέλη. Για παράδειγμα, έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα από τα Ταμεία Life για να βελτιωθεί η κατάσταση. Νομίζω στη Γερμανία είναι αυτό, αλλά τα καλά αποτελέσματα θα διαδοθούν προσπαθούμε να ε, δώσουμε και την ευκαιρία στους πολίτες να χειραφετηθούν και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους αλλά και ε, η αποτελεσματικότητα που καμιά φορά σε εθνικό επίπεδο χρειάζεται λιγότερος χρόνος από ό,τι σε ευρωπαϊκό για να ε, εκδοθεί μια δικαστική απόφαση. Και τα κρατη με έλαβαν μέτρα αφού έχουμε προσφυγή εις βάρος τους επί δεν είναι πολύ εύκολο να αλλάξουν όμως κάποιες δομές και κάποιες πρακτικές. Γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια σε κάποια κράτη-μέλη που χρειάζεται να αλλάξει τελείω ο τρόπος ζωής μας. Είναι η θέρμανση των κατοικιών στην Ανατολική Ευρώπη, είναι η κυκλοφορία, είναι οι μεταφορές, είναι συγκοινωνίες καμιά φορά και οι κλιματικές συνθήκες ας πούμε στην κοιλάδα του Πάδου στην Ιταλία και το, το ανάγλυφο ε, του εδάφους, η μορφολογία κτλ. Ε, για τον έλεγχο τώρα και την παρακολούθηση θέλω μόνο να προσθέσω ότι από νομική σκοπιά πάλι το εξετάζουμε και έχουμε και αμφισβητήσεις για το πώς μετράνε κάποια κράτη-μέλη. Στο Βέλγιο έχουμε αυτή την ανησυχία για τον έλεγχο και την παρακολούθηση και για το σημείο μέτρησης αγλουά. Πάντως το βλέπουμε ευρύτερα, έτσι, τη συνολική εικόνα για το τι σημαίνει στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και ε, μέσα που διαθέτουμε και οι δυνατότητες μας έχουν και τα όρια τους. Ε, κάποια πρόοδο τη βλέπουμε όμως στα κράτη-μέλη, ό,τι και να πούμε. και τα πιέζουμε, δεν τα αφήνουμε έτσι ελεύθερα. Ευχαριστώ. Άντε παιδί, σφύρα το. Uh, uh, Πάρα πολύ χρήσιμη η συζήτηση. Τώρα θα κηρύξω το πέρα συνεδρίαση. Η επόμενη συνεδρίαση δε, δεν έχουμε και διάφορα, θα είναι 7 και 8 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ. Τα λέμε.